So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα την εντύπωση ότι δεν είχαμε χρησιμοποιήσει σωστά τα μέσα επικοινωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο για να επικοινωνήσουν οι επιτροπές. Έχουν περιορισμένο χρόνο όμως. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε την κοινή αυτή ακρόαση Επιτροπής ΕΚΟΝ και Επιτροπής Απασχόλησης για λόγους, συνέπειες και διόρθωση των οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω τους αγορητές που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Ξεκινώ με τη σειρά που θα μιλήσουν. Δεν έχει σχέση με την αλφαβητική σειρά. Ο κ. Μακφέρσον από τον ΟΣΑ, υποδιευθυντής για θέματα απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων και εργασία Η κυρία Κέιτ Πικέτ, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του York και ο κ. Μάρκ Τεφώση, καθηγητής Ευρωπαϊκής και διεθνού Απασχόλησης και Εργατικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Γάνδη. Σα ευχαριστώ πολύ. Καταφτάσατε εγκαίρω. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ίσως το γνωρίζετε ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και οι σχετικές πολιτικές απαντήσεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις ανισότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αύξησαν σημαντικά ε, ε, το ξέσπασμα αυτό και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Η αύξηση των ισοτήτων επηρεάζει την αντίληψη που έχουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις λύσεις που περιμένουν από τους νομοθέτες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η ΕΚΟΝ και η ΕΜΠΛ που ζήτησε να συμμετάσχει στη διοργάνωση ακρόασης λόγω των ενισοτήτων εξετάζουν και δύο επιτροπές, λέγω γι' αυτό πρέπει να εστιαστούν επί των οικονομικών ανισοτήτων και τι συνέπειε έχει αυτό για την ανάπτυξη και για τις λύσεις των προβλημάτων. Καλωσορίζω λοιπόν του ομιλητέ μας. Τους δίνω τη σειρά, με τη σειρά που προανέφερα το λόγο. Ο κ. Μακφέρσον λοιπόν είναι ο πρώτο ο οποίο θα λάβει το λόγο. Υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, είμαι από το Κέντρο ε, Ευκαιριών και απασχόληση στο ΩΣΑ και θα μιλήσω για τις ανισότητες τις ισοδηματικές. Όχι διότι είναι πιο σημαντικές οι ισοδηματικές ανισότητες από τις πτυχές κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά είναι καλύτερα τεκμηριωμένη αυτή η ισότηση. Αν ε, συνεχίσουμε, γιατί τεκμηριώνεται καλύτερα, πάμε στην αρχή της δεκαετίας του 90, κατέληξαν πολλές προσπάθειες να τυποποιήσουμε το πώς προσμετρούμε τις ανισότητες στις διάφορες χώρες και επίσης σειρά ετών μετά εκπονήσαμε στατιστικά στοιχεία πολλά για την ανισότητα και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε, για να το πω ειλικρινά. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε μέχρι ότου φτάσουμε στο τέλος της δεκαετίας του 2000, 2008 περίπου, όπου επιτέλους δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή, επιτέλους τη σημασία που έχουν οι ενισότητες και έγινε κατανοητή η ταχεία αύξηση των ενισοτήτων επί μακρά περίοδο. Στην επόμενη διαφάνεια ε, βλέπετε τα παρόντα επίπεδα ανισοτήτων έχουμε έναν ε, ε, συντελεστή που δεν μπορούμε να τον ε, παρουσιάσουμε. Κάτι σαν τη θερμοκρασία είναι. Το συντελεστή Gini περίπου 25 είναι αρκετά ευχάριστα τα πράγματα. Άμα πα στα 30, κάπω ζεσταίνεσαι και όταν φτάσει στα 35 ή στα 40, αισθάνεσαι δυσάρεστα. Είναι ένας καλός τρόπος να βλέπει κανείς τα επίπεδα ανισότητα. Αν βλέπετε το γράφημα, έχουμε Ευρωπαϊκές και σκανδιναβικές χώρες που έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα ανισοτήτων και εντό της Ευρώπης ε, οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ανισοτήτων ε, αλλά είναι σημαντικά κατώτερα αυτά τα επίπεδα από ό,τι βλέπει κανείς εντός Ευρώπης. Ε, το σημαντικό είναι ότι οι ενισότητες ε, αυξάνονται επί μακρά χρονική περίοδο, σχεδόν σε κάθε χώρα. Ναι, υπάρχουν κάποιες χώρες εκεί που δείχνουν μια κάποια σταθερότητα. Στην τεράστια όμως πλειοψηφία των χωρών βλέπετε σημαντικές αυξήσεις ανισοτήτων για να το πω διαφορετικά, από το 1985 και μετά τα εισοδήματα του πάνω 10% αυξήθηκε περίπου 55% σε πραγματικούς όρους, τα εισοδήματα του κάτω 10% αυξήθηκε περίπου 15, 10 με 15% σε πραγματικούς όρους. Είναι να το πούμε διαφορετικά, τα μέσα της δεκαετίας του 80 το ποσοστό εισοδημάτων του πλουσιωτέρου 10% προς το 10% φτωχότερο ήταν 7 προς 1. 7 φορές παραπάνω είχαν οι πλουσιότερες φτωχότερες. Τώρα 10 φορές παραπάνω δεν είναι μικρή αύξηση στην ανισότητα. Δεν θα έχω χρόνο να πω πολλά για τη φτώχεια, αλλά και αυτό είναι απίστευτα σημαντικό δεν είναι το ότι η φτώχεια απλώς αυξήθηκε. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, δεν μπορούμε να πούμε τι έγινε με τη φτώχεια, αλλά εκείνη που είναι φτωχοί σίγουρα έχει αλλάξει η κατάστασή του. Τα μέσα της δεκαετίας του 80, αν ήσουν πάνω από 75, ήσουν δύο φορές περισσότερο πιθανό να είσαι φτωχό από το μέσο άνθρωπο, τον πληθυσμό. Τώρα γνωρίζεις περισσότερο. Δεν, είσαι, δεν είναι τόσο πιο πιθανό να είσαι πιο φτωχό στον υπόλοιπο πληθυσμό. Έχει αλλάξει το πράγμα πολύ μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τα επίπεδα της φτώχειας ή τις πιθανότητες να είναι κάποιος φτωχός αν είναι ηλικιωμένος. Αντίθετα, εκείνοι που είναι πολύ πιθανότερο να είναι φτωχότεροι από ό,τι ήταν πριν οι με παιδιά και οι νέοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε γιατί μας νοιάζει τόσο πολύ αυτή η ανισότητα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς το να είναι φτωχός όταν έχει παιδιά έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες πολύ πιο μεγάλες και έχει και αντίκτυπο στην οικονομική υγεία της χώρας. Ε, νομίζω ότι βλέπουμε στην επόμενη διαφάνεια, προχωρώ μέχρι ότου να καλύψουμε όλα τα τετραγωνάκια. Γιατί η ανισότητα αυξάνεται. Ε, βλέπουμε διάφορους παράγοντες. Λοιπόν, πρώτο σημαντικός προφανής παράγων είναι η αλλαγή στην απασχόληση. Ε, κάποιοι είναι πολύ πιο πιθανό να βρουν δουλειά, να εργαστούν και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες. Ε, ε κυρίως έχουμε αύξηση στις άτυπες μορφές ε, εργασίας, προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση. Έπαιξαν σημαντικό παράγοντα ισότητας. Δεύτερος παράγοντας, η ανακατανομή είναι λιγότερο αποτελεσματική. Δεν είναι ότι δαπανούμε λιγότερα όσον αφορά τα συστήματα, τα ανταποδοτικά κλπ αλλά ξοδεύουν περισσότερα. Αλλά ο τρόπος που έχουμε φορολόγησης ε, και ευεργετημάτων κάνει χειρότερη ανακατανομή. Δεν τα πάμε τόσο καλά πια να παίρνουμε του πλούσιου και ανήμου φτωχού. Και τρίτο σημαντικό παράγονο είναι οι τεχνολογικέ αλλαγέ που βασίζονται στι δεξιότητε. Η φύση των τεχνολογικών αλλαγών που επιβραβεύει εκείνους που έχουν δεξιότητες περισσότερο από εκείνους που δεν έχουν δεξιότητες. Και είναι μια βαθιά υποβόσκουσα τάση και είναι πολύ δύσκολο οι νομοθέτες να αντιδράσουν σε αυτό, αλλά είναι ένας βασικούς λόγους για τους οποίους είδαμε αύξηση της ανισότητας με τον βάρο του χρόνου. Και υπάρχει και αυτό που βλέπουμε μετά τα τραγωνίδια διακεκομένες γραμμές. Έχουμε πιο πολλές μονογαμικές οικογένειες Έχουμε επίση παρόμοιους, κοινωνικών τάξεων ανθρώπου να πατρεύονται. Άλλαξε η μορφή των γάμων και των οικογενειών. Μετά υπήρχαν και κάποιε αντισταθμιστικές συνέπειε. Πρώτα απ' όλα έχουμε την αύξηση τη παιδεία, τη εκπαίδευση, ε, που εξισώνει τα πράγματα, η παιδεία, όσο καλύτερα τα καταφέρνεις να παραμένουν στην παιδεία επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο μειώνει τι ανισότητε σε μεταγενέστερο στάδιο τη ζωή του. Δεύτερο σημαντικό παράγον που δεν είναι γνωστό είναι οι γυναίκε. Όλο και περισσότερε γυναίκε ε, εργάζονται και μειώνεται επίση και η ανισότητα των αμοιβών λόγω φύλου, η έμφυλη διαφορά. Έχουμε δρόμο να κάνουμε, παρόλα αυτά οι ανισοτητε γενικά έχουν μειωθεί. Ε, κυρίως η ανισότητα που θα αυξανόταν 5% παραπάνω από ό,τι έγινε από τα μέσα τη δεκαετία του 80 αν οι γυναίκες ακόμα συμπεριφερόταν με τον τρόπο που συμπεριφερόταν κατά το παρελθόν, αν εργαζόταν λιγότερο ή να αμοιβόταν λιγότερο όπως τα μέσα της δεκαετίας 80. Περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας ε, ε, ξισώνει τα πράγματα όσον αφορά την οικονομία μας. Τώρα θα ήθελα ακροθυγώς να αναφερθώ στα, σε συνέπειες των μεγαλύτερων ισοτήτων. Βέβαια υπάρχουν κοινωνικοί αντίκτυποι, πολιτικοί αντίκτυποι, υπάρχουν εντολικοί λόγοι για τους οποίους μας νοιάζει η ανισότητα Είμαι οικονομολόγος, εγώ συσταθώ επί των οικονομικών αντικτύπων των ανισοτήτων. Ε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στις οικονομίες και πρέπει να το λησμονούμε μετά. Ε, όταν ε, ψάξουμε βλέπουμε ότι οι οικονομίες που έχουν μεγαλύτερε ανισότητες έχουν χαμηλότερη ανάπτυξη και είναι σχέση αιτίου αιτιατού. Όσο αυξάνεται η ανισότητα, έτσι πιστεύουμε ότι και η ανάπτυξη μειώνεται Εξήγησα εδώ ότι μια αύξηση στην ανισότητα κατά ένα σημείο τζίνι μειώνει κατά 0,1 την ανάπτυξη ε, το χρόνο. Δηλαδή η αύξηση της ανισότητας που έδειξα πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έχει συνεπιφέρει περίπου, έχει αφαιρέσει 5% περίπου ε, την αύξηση του εισοδήματος. Είναι σημαντικό αποτέλεσμα που έχει ανισότητα όσον αφορά την ανάπτυξη. Τώρα γιατί διότι καταρχάς το σημαντικότερο είναι κάτι που δεν σχετίζεται με τη φτώχεια, αλλά σχετίζεται με όλους που είναι στο κάτω τμήμα της κοινωνίας, το 40%. Με μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του χαμηλού 40% και των υπολείπων, τόσο πιο αρνητική συνέπεια στην ανάπτυξη. Και αυτό σχετίζεται με πράγματα που υποψιαζόμαστε όπως είναι η υγεία, όπως οι κοινωνικές επαφές, αλλά αυτό που καταφέραμε πραγματικά να εντοπίσουμε είναι η παιδεία. Προφανώς οι φτωχοί άνθρωποι είναι πολύ λιγότερο πιθανό να είναι στην παιδεία από ότι πλούσιοι. Αλλά ακόμα και αν διατηρήσει σταθερό το επίπεδο του εισοδήματο, όσο αυξάνεται η ανισότητα στην κοινωνία, τόσο οι πιθανότητε ο κόσμο να εκπαιδεύεται. Και όσο πιο χαμηλή και η πιο χαμηλή ποιότητα της παιδείας που δέχονται. Αυτά μαζί έχουν συνεχή αποτελέσματα όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο στην οικονομία και το ρυθμό ανάπτυξη οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο είναι ο βασικό λόγος για τον οποίο η ισότητα επηρεάζει τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Επίσης εκεί δείχνουμε ότι η ανακατανομή ε, δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στι αναπτυγμένε χώρε. Διαφορετικά στι αναπτυσσόμενε χώρε. Στι αναπτυσσόμενε χώρε δεν έχουμε στοιχείο ότι η μεγαλύτερη ανακατανομή είναι κάτι κακό για τα επίπεδα τη ανάπτυξη. Τελευταίο που έχω να πω για διευθυντικά μέτρα, διότι αυτό ήταν και ο τη της σα. Έχουμε τέσσερις τομείς που εξετάζουμε, πολλοί από αυτούς δεν θα σα εκπλήσουν. Πρώτα απ' όλα απασχόληση, αλλά όχι απλή απασχόληση, σε πολλέ χώρες προσωρινή απασχόληση, άτυπε μορφέ εργασία είναι παγίδα. Δεν είναι εφαλτήριο, είναι παγίδα, οπότε δίνουν μόνιμα κακέ θέσει εργασία. Θα πρέπει ο κόσμο να κάνει καριέρα, όχι μόνο να μπαίνει σε οποιαδήποτε προσωρινή δουλειά ή άτυπη μορφή εργασία. Το δεύτερο που συνεπάγεται από τα προλαλήσαντα, αυτά που προαναφέραμε, όσο περισσότερε γυναίκε μπαίνουν σε θέσει εργασία και όσο πιο πολύ μπορούμε να μειώσουμε τι διαφορέ αμοιβών ανδρών και γυναικών, τόσο τα καλύτερα θα τα καταφέρνουμε για τη μείωση των ισοτήτων. Τρίτο, προφανέστατο βεβαίω, πρέπει να ενισχύσουμε την παιδεία και τις δεξιότητες και τέταρτον ε, που θέλω να αναφέρω είναι να πω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα ή τουλάχιστον κάποιε χώρε στην Ευρώπη μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα όσον αφορά τη βελτίωση σχεδιασμού του συστήματο φορολόγηση και βεγεδημάτων για να μειωθούν οι ανισότητε χωρί να αυξήσουν απαραίτητα τι δημόσιε δαπανών, έχοντα συγκεκριμένη στόχευση όσον αφορά του φόρου και τα ευεργετήματα για να μειωθούν οι ανισότητε. Εν συντομία, αυτή ήταν η παρουσίασή μου και προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Πικέτη, η δεύτερη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας εξηγήσω ποιες είναι οι επιπτώσεις αλλά και τα μέτρα διόρθωσης που θα μπορούσαμε να είχαμε για την οικονομική ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά μιλάω στους πολίτες, στο κοινό, για όλη αυτή την έρευνα, την ποσοτική έρευνα που έχει γίνει όσον αφορά το φαινόμενο αυτό. Αν καταλάβετε αυτή τη γραφική παράσταση, πραγματικά τα καταλαβαίνετε όλα. Η ανισότητα αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τον κόσμο όπως προέκυψε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση των προηγούμενων ετών και πλήττει τόσο πλούσιες όσο και φτωχές χώρες. Οι ανισότητες δημιουργούν οικονομική αστάθεια, όπως ακούσαμε, καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό, υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, καταστρέφουν την υγεία των πολιτών και δεν επιτρέπουν την έγκριση στρατηγικών που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η κοινωνική και οικονομική λοιπόν ανισότητα δεν επιτρέπει στα άτομα και στις κοινότητες να φτάσουν σε ένα καθεστώς ευημερίας, να κμάσουν και ουσιαστικά δημιουργούν πάρα πολλούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και όσο κατεβαίνουμε στα πιο χαμηλά οικονομικά κοινωνικά στρώματα, τόσο περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουμε και τόσο μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ φτωχών και πλούσιων μολονότι οι επιπτώσεις της ανισότητας φαίνεται να είναι περισσότερες για τους πιο φτωχούς, ακόμα και οι πιο πλούσιες χώρες και τα πιο πλούσια κοινωνικά στρώματα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λόγω της ανισότητας. Έχουμε πολλές φορές συνταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων για αυξημένα επίπεδα άγχους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί στα πλαίσια μιας κοινωνίας που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ε, ανισότητας και δεν καταφέρνουμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταλήξουμε σε πιο ισότιμες κοινωνίες. Και α μην ξεχνάμε πολλέ φορέ ότι υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στα κοινωνικά και υγειονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι χώρε, αλλά τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται πολύ περισσότερο στι χώρε εκείνε οι οποίε πλήττονται από οικονομικά προβλήματα και από αυξημένα προβλήματα ανισότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα κάποιους δείκτες όπως το κατακεφαλή ΝΑΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί λοιπόν η ανισότητα προκειμένου να αυξηθεί η ευημερία των πολιτών. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ότι αυτές οι πολύ μεγάλες διαφορές οι κοινωνικές είναι ιδιαίτερα επιζήμιες. Ας δούμε την προηγούμενη διαφάνεια. Η ανισότητα επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής, αυξάνει την θνησιμότητα. Επίσης έχουμε θνησιμότητα των παιδιών, ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία είναι υψηλότερα στις πιο άνισες κοινωνίες. Επίσης αυξάνονται τα επίπεδα του AIDS και του μόλυνση, της μόλυνσης από το HIV. Επηρεάζονται επίσης οι κοινωνικές ε, σχέσεις. Η κοινωνική συνοχή πλήττεται το ζήτημα της ε, εμπιστοσύνης. Κάποιοι δείκτες που έχουν να κάνουν με το καθεστώς των γυναικών είναι καλύτεροι στις πιο ισότιμες ε, κοινωνίες, ενώ στις κοινωνίες που παρουσιάζουν μεγάλα επίπεδα ανισότητας εμφανίζονται και μεγαλύτερα προβλήματα εγκληματικότητας ή όπως ανθρωποκτονίες λοιπά. Επίσης επηρεάζονται ακόμα και οι ευκαιρίες που έχουν τα ίδια τα παιδιά. Σύμφωνα με την UNICEF, η ευημερία των παιδιών είναι σαφώς υψηλότερη σε χώρες οι οποίες, ή σε κοινωνίες που είναι πιο ίσες. Αντίθετα, στις κοινωνίες εκείνες που πλήττονται από ανισότητα έχουμε περισσότερα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο και περισσότερες ε, κοπέλες ε, οι οποίες αποκτούν παιδιά την, εποχή της, την περίοδο της εφηβείας είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι λόγω της ανισότητας επηρεάζονται και ίσες ευκαιρίες, οι οποίες προφανώς μειώνονται. Δεν είναι μόνο υγειονομικά τα προβλήματα, τα κοινωνικά τα προβλήματα προκαλεί ανισότητα, όπως είπε ο Μάρκα πριν από λίγο, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε τους τρόπους με τους οποίους η ανισότητα επηρεάζει την οικονομική σταθερότητα και την πρόοδο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι, ακόμα και βραβευμένοι με το Νόμπελ Οικονομίας, οι οποίοι συμφωνούν με την προσέγγιση αυτή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας λέει ότι η μείωση της ανισότητας και αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματο. Επίση, η ανισότητα συνδέεται με μικρότερες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργεί πιο έντονους ε, οικονομικούς κύκλους που παρουσιάζουν ακραίες τάσεις, δηλαδή είτε απότομη και σύντομη οικονομική ανάπτυξη που συνοδεύεται από περίοδους ύφεση. Όλο και περισσότερο οι ηγέτες ασχολούνται περισσότερο με την ανισότητα και αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι η ανισότητα πραγματικά δεν μας βοηθά να καταλήξουμε σε μια πιο σταθερή οικονομία. Ακριβώς επειδή δημιουργεί εσωτερικούς ανταγωνισμούς, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες τάσεις για ορισμένες κοινωνικές ομάδες όσον αφορά τον καταλωτισμό. Συντοποιούμε ότι ε, οι ε, κοινωνίε οι οποίε δεν έχουν προβλήματα ανισότητα λειτουργούν πολύ καλύτερα, πολύ πιο επεύθυνα από οικονομική πλευρά. Συντοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι ε, σε κοινωνίε που δεν πλήττονται από ανισότητα τηρούνται καλύτερα και διάφορε διεθνεί συμφωνίε όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Ο δέκατο στόχο των παγκόσμιων στόχων ανάπτυξης έχει ως στόχο τη μείωση της ανισότητας ανάμεσα στις χώρες και ο στόχος 10.1 είναι ότι μέχρι το 2030 να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα ενισχυμένο εισόδημα για το 40% του πληθυσμού που βρίσκεται στο χαμηλότερο οικονομικό εισοδηματικό επίπεδο. Μόνο αν καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την ισότητα, θα έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη σε πλούσιες και φτωχές χώρες, η οποία δεν θα δημιουργεί αποκλεισμούς και θα οδηγεί στην ευημερία των πολιτών. Οι εισοδηματικές αυτές διαφορές μπορούν να μειωθούν κατά δύο τρόπους, μέσω της ανακατανομής, μέσω των φόρων και των επιδομάτων, είτε με την εξισορρόπηση των εισοδημάτων πριν την καταβολή των φόρων. Στην έρευνα που έχω κάνει μαζί με άλλους ερευνητές, βλέπουμε ότι και οι δύο αυτές μέθοδοι συμβάλλουν τελικά στη μείωση της ανισότητας εξίσου. Δεν έχει μεγάλη σημασία ποια μέθοδο ακολουθεί κανείς, αρκεί να φτάσει στο ευκταίο αυτό αποτέλεσμα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι πιο αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, η αντιμετώπιση όμως των φορολογικών παραδείσεων, η καλύτερη ανακατανομή του πλούτου, η πιο υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων είναι καθοριστική σημασία ζητήματα, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της διεθνού συνεργασίας. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή όχι μόνο δημιουργεί μεγαλύτερη ανισότητα, αλλά ένα πολύ μεγάλο τμήμα των χρημάτων που θα πήγαιναν στον κρατικό προπολογισμό πρέπει αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτηθούν τελικά από τους πόρους που έχουν τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Προφανώς κάτι τέτοιο πρέπει να αλλάξει. Αλλά μπορεί να ριζωθεί με ένα καλύτερο τρόπο η αντιμετώπιση της ανισότητας στα δημοκρατικά πολιτεύματα εις όλες τις κοινωνίες και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της καλύτερης συνεργασίας, της πιο υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Ξέρετε ότι στην Ισπανία υπάρχει μια οργάνωση ε, εργοδοτών που ε, απασχολεί 80.000 ανθρώπους και ο λόγος εδώ εισοδηματικής διαφοράς είναι 15 προς 1. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια πιο, μια πιο δίκαιη βάση προκειμένου να μπορούν όλοι οι πολίτες να λειτουργούν και να ζουν ισότιμα. Αν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, και το τονίζω αυτό, είναι αποδεικτικά στοιχεία, είναι νέα για εσά, τότε μπορείτε να πάτε σε αυτή την ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερε πληροφορίε αλλά και επικαιροποιήσει των ερευνών αυτών. Είτε είναι νέα τα στοιχεία αυτά, είτε είναι ήδη γνωστά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσετε την αντιμετώπιση τη ανισότητα στο κέντρο των πολιτικών και τη στρατηγική σα είναι ο καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου όλε οι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσουν το βιωτικό επίπεδο, την ευμερία όλων των πολιτών, να σταθεροποιήσουν την οικονομία και να οδηγηθούν προ τη βιωσιμότητα. Κατάφεραν στα πόλα σε 7,5 λεπτά. Σα ευχαριστώ. Thank um, ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω τώρα τον λόγο στον κύριο Μάρκ Ντεφό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μου δίνετε 10 λεπτά για να αναφερθώ σε ένα από τα πιο περιπλοκά ζητήματα του καιρού μας. Θα ξεκινήσω με την πρώτη διαφάνεια. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω τα όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, να δώσω κάποιες επιπλέον πρόπτικες. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Μάρκ, θα ήθελα λίγο να πω κάποια πράγματα η περίοδος αναφοράς που χρησιμοποιούν όλοι, ρητός ή όχι, συγκρίνει τα όσα ζούμε σήμερα με την περίοδο που σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 που ήταν ένα χαμηλό ιστορικό ανισότητας. Είναι μια ιστορική ανομαλία ίσως, αλλά τουλάχιστον ήταν ένα ιστορικό χαμηλό. Καλό είναι να το θυμόμαστε όταν κάνουμε σύγκριση σε αυτό το οποίο άλλαξε στον κόσμο μεταξύ τότε και τώρα είναι αρκετά πράγματα. Θα ήθελα να τονίσω πως η αυξανόμενη ανισότητα, η οικονομική ανισότητα, ειδικά του εισοδήματος, είναι αντικατοπτρισμός ενός προβλήματος οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αυτή που ήταν όσον αφορά την ε, ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας και δεν το συνειδητοποίησαμε γρήγορα γιατί είχαμε κρύψει κάτω από το χρέος ε, την μη αύξηση της παραγωγικότητας αλλά αυτό το ανέδειξε η ε, κρίση του χρέους. Οπότε τα ζητήματα της παραγωγικότητας προϋπήρχαν ε, της αύξησης της ανισότητας. Δεύτερον, πρόκειται για ένα φαινόμενο της ανάπτυξης, γιατί έχουμε τομείς νέας ανάπτυξης, εντυπωσιακής μάλιστα, και μάλιστα από κλάδους ε, που δημιουργούν τρομερή συγκέντρωση ε, εισοδήματο και όχι διανομή του. Μιλάμε για την τεχνολογία, τη χρήση του διαδικτύου, την παγκοσμιοποίηση και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ειδικευμένοι και μπορούν έτσι να κερδίσουν πάρα πολλά σε μια παγκόσμια αγορά. Σχεδόν οποιοδήποτε στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος είναι επιτυχημένος σήμερα στην Δύση ε, κερδίζει λεφτά εκτός της χώρας του λόγω της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Οπότε οι δυνατότητες του είναι πολύ υψηλότερες και δεν είναι πλέον εθνικές εγχώριες σε σύγκριση με άλλα άτομα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με αυτό το ευρύτερο κύμα θα λέγαμε οικονομικής ανάπτυξης. Οπότε υπάρχει ένα φαινόμενο ανάπτυξης με την έννοια ότι σε σύγκριση με το παρελθόν με την περίοδο που τελείωσε το 1970 και ξεκίνησε με την άνοδο μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Δεν μπορούν τώρα όλοι να υποφεληθούν με τον ίδιο τρόπο όπως ε, στο παρελθόν στην περίοδο της ανοικοδόμησης. Αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό, αλλά είναι σαν τον καιρό. Δηλαδή μπορούμε να παραπονιόμαστε, αλλά είναι δύσκολο να αλλάξει εκτός εάν ε, γίνουν παγκόσμι, εκτός αν παγκόσμιες αλλαγές. Οπότε, αν κοιτάμε την ανισότητα σε οποιαδήποτε κλίμακα, θα δούμε μεγάλες διαφορές μεταξύ κλάδων της οικονομίας ε, αν συγκρίνουμε εταιρείε εντός ενός κλάδου και αν συγκρίνουμε άτομα εντός εταιρείων. Παραδείγματος χάρη μιλάμε για την γνώση και ο συνάδελφος είπε πως ε, η εκπαίδευση εξισώνει ως ένα βαθμό αλλά ταυτόχρονα πολλώνει κιόλα γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, υψηλή εκπαίδευση και μόρφωση μπορούν τώρα να έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες εσόδων από ό,τι στο παρελθόν και βλέπετε ότι δίνει ευκαιρία σε άτομα ε, αντί να εξισώνει αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ πέρα ανησυχητικά. Μιλάμε για την ανισότητα με βάση ένα μοντέλο συνένεση σε όλες σχεδόν τις ε, δυτικές δημοκρατίες, δηλαδή θεωρούμε την αγορά το μέρος το οποίο δημιουργείται η ευημερία και ελέγχεται από το κράτο και τα όσα παράγει η αγορά μετά χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί ένα κράτο πρόνοια. κάπω έτσι τα βλέπουμε. Από αυτή την σκοπιά λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε ερωτήσει και πολλοί έχουν κάνει ερωτήσει και ο Στίγκλιτ που αναφέρθηκε για το εάν η αγορά είναι ακόμα αγορά. Αν δούμε παραδείγματο χάρη τα φαινόμενα συγκέντρωση του διαδικτύου με τις πλατφόρμε, τα φαινόμενα του ε, δικτύου, με την παγκοσμιοποίηση. Βλέπουμε λιγότερο ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι θετικό εάν θεωρούμε πως η ε, ανισότητα είναι κάτι το οποίο κερδίζει κανείς ή αξίζει κανείς χάρη στην απόδοσή του. Και συμπληρωματικό προς αυτό υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο το οποίο συχνά αγνοούμε είναι ότι πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας ε, της τελευταία δεκαετία έχουν πάει στον μη κερδοσκοπικό τομέα Εκπαίδευση δηλαδή, υγεία και ανάλογες τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό είναι, ισχύει και στη χώρα μου. Βέλγος είμαι. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Αν είναι κανείς δάσκαλος, γιατρός, νοσοκόμος και θέλει να αυξήσει τα έσοδά του, πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητα. Αυξημένη παραγωγικότητα σημαίνει ότι ο δάσκαλος θα διδάσκει λιγότερο. Ο νοσοκόμος θα νοσηλεύει λιγότερο ή θα πει εάν είναι να επενδύσω σε σένα και θα γίνεις πιο παραγωγικός μου κοστίζεις περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσει περισσότερα το κράτος γιατί το κράτος επιδοτεί. Οπότε ξεκινάμε αυτό το οποίο λέγεται η ασθένεια του κόστους, δηλαδή ένας μεγάλος κλάδος της οικονομίας. Δεν μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα χωρίς να επηρεάσει το κόστος για τον καταναλωτή ή την ποιότητά του. Οπότε έχουμε μια πρόκληση στις κοινωνίες της δύση και βεβαίως όσο η κοινωνία γυράσκει, οι κλάδοι αυτοί αυξάνονται. Θα πείτε ότι έχουμε μια λύση. Ναι, βεβαίως υπάρχει λύση. Να προσθέσουμε την τεχνολογία στην εξίσωση. Τι σημαίνει αυτό, λιγότερους γιατρούς, λιγότερους νοσηλευτές, ε, λιγότερους δασκάλους. Και έχουμε μετά ξανά αυξημένη πόλωση. Οπότε έχουμε... είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δεν είναι εύκολο να βγει κανεί ε, χωρίς κάποια ανάπτυξη σε άλλους κλάδους οικονομίας. Ένας άλλος μεγάλος τομέας για τα τελευταία 40 χρόνια είναι αυτό το οποίο ο Μπεν Μπερνάνκε πριν από την μεγάλη κρίση έλεγε την ε, μεγάλη μετριοπάθεια, δηλαδή ότι οι κεντρικές ε, τράπεζες είχαν καταφέρει λίγο πολύ να ελέγξουν τις διακυμάνσεις του καπιταλισμού και είχαμε λιγότερε κρίσεις από ό,τι είχαμε ιστορικά. Και είναι σημαντικό να έχουμε ε, κατά μια ιστορική προοπτική. Οπότε έχουμε πράγματι ε, μέχρι στιγμή ένα θετικό ιστορικό αύξησης ε, των θέσεων εργασία και υπάρχουν αυτά στη σχετική βιβλιογραφία και ο Μπεν Μπερνάγκη τα χειράψε, αλλά υπάρχει και η άλλη πτυχή Δηλαδή αν υπάρχει σταθερότητα στις χρηματαγορές και χρησιμοποιούμε τα λεφτά για να απαλύνουμε τους κύκλους της οικονομίας, δημιουργούμε ένα κλάδο ο οποίος ε, κινείται από το χρέος και γι' αυτό έχουμε δει ακριβώ μια αύξηση, μια αύξηση των επιπέδων χρέους ε, και βεβαίω ε, τη χρηματοπιστωτική οικονομία. Γι' αυτό όσοι μπορούν να επενδύσουν σε αυτά έχουν μεγαλύτερο κέρδο και όσοι έχουν διαθέσιμο κεφάλαιο μπορούν να το επενδύσουν ή να αποκτήσουν ακόμη περισσότερο κεφάλαιο. Οπότε η αποκτησουν ακομη περισσοτερο κεφαλαιο πτυχή τη σταθεροποίηση έχουμε τη σταθερότητα και δημιουργία θέσεων εργασία, αλλά έχει και την άλλη όψη τη ανισότητα που βασίζεται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Δεν σταματάει εύκολα αυτό αν το κάνει αν το κάνουμε ήδη εδώ και πάνω από 30 χρόνια, όπως το κάνουμε, και δεν το σταματήσαμε. Είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε λοιπόν να αναφερθούμε στην κρίση του ευρώ, η οποία δεν έχει τελειώσει. Γίνεται μία διαχείριση, αλλά δεν έχει επιληθεί. Πώς την διαχειριζόμαστε, κυρίως βασιζόμαστε ξανά σε νομισματική πολιτική, ξανά το ίδιο πράγμα κάνουμε. Οθούμε τις χρηματαγορές για να επενδύσουν αυτοί που έχουν λεφτά και τιμωρούμε αυτούς που έχουν μόνο λεφτά να αποταμιεύσουν και δεν μπορούν να επενδύσουν. Αυτό είναι η παρενέργεια μιας πολιτικής, η οποία είναι αναγκαία πολιτική, εάν δεν υπάρχει μια αναλλακτική μακροοικονομική πολιτική, βεβαίω στρεφόμαστε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Τι πέρασε ο χρόνος μου, μάλιστα. Λοιπόν, πόλωση, λοιπόν, αυτό συμβολίζει αυτή η εικόνα. Λοιπόν, Όταν μιλάμε για ανισότητα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους ε, τρόπους. Η δυσκολία με τα στατιστικά στοιχεία της ανισότητας είναι ότι έχουν μία τάση να είναι συνολικά στατιστικά. Δηλαδή, αν πάμε πέρα από τα ε, στατιστικά σε επίπεδο χώρας, όπως ο συντελεστής ε, Τζίνι, βλέπουμε διαφοροποίησεις. Δεν λέω πώ δεν αυξάνεται δηλαδή η ανισότητα, αλλά είναι κάπως πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Παραδείγματος χάρη, η παγκοσμιοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μειώσει την ανισότητα μεταξύ χωρών. Είναι η τάση γενική. Υπάρχουν εξαιρέσει, αλλά η τάση γενική είναι αυτή. Δηλαδή, έχει αυξηθεί η ανισότητα εντό τη Δύση, όπου έχει χαθεί κάποια δυνατότητα στη βιομηχανική παραγωγή γιατί παράγουμε στην Κίνα, αλλά αυτή η ανισότητα στην Δύση αντικατοπτρίζει την μέση τάξη που δημιουργήθηκε στην Κίνα. Και σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει μείωση στην ανισότητα μεταξύ χωρών. Δεύτερον, αν δούμε τις χώρες. Βεβαίως οι χώρες μπορούν να έχουν μεγάλες εσωτερικές διαφορές. Αν δείτε τη χώρα μου, το Βέλγιο, και δείτε τα στατιστικά στοιχεία του συντελεστή Τζίνι θα δείτε ότι το Βέλγιο δεν τα πάει άσχημα. Δεν, δεν υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Μα εξαρτάται. Αν ζει κανεί στο νότο τη ε, χώρα, η πραγματικότητά του είναι διαφορετική από ό,τι στο βορρά. Αν ζει κανεί στι ε, Βρυξέλλε και είναι μετανάστη, είναι τελείω διαφορετική ε, από ότι αν ζει στη Δυτική Φλάνδρα όπου υπάρχει πλήρη απασχόληση. Ε, Τεράστιε διαφορέ και στι ΗΠΑ και αλλού. Υπάρχουν μεγαλοπόλει, ε, μεγάλε πόλει που είναι πολύ άνισα μέρη και η πραγματικότητα βεβαίω εκεί πέρα είναι διαφορετική από ό,τι στην Ήπεθρο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί πριν ε, φτάσουμε βιαστικά σε συμπεράσματα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο έργο του Πάτναμ εδώ πέρα, ε, πρωτοπόρος της Ήπα. Ε, εντός της ίδιας χώρας, και το ανέφερα ήδη και θα σταματήσω, εντός της ίδιας χώρας βλέπουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ ε, κοινωνικών και εθνοτικών μάθων. Αυτό σχετίζεται εν μέρη με την χειραφέτηση των γυναικών και το τι γίνεται εντό των οικογενειών, γιατί μετράμε κυρίως με την οικογένεια ως μονάδα. Οπότε η χειραφέτηση σημαίνει λιγότερη ανισότητα μεταξύ των φίλων και περισσότερη ανισότητα μεταξύ των οικογενειών. Και ε, βεβαίω υπάρχουν και οι ήρωές τη μετανάστευση που έχουμε από την δεκαετία του 1970. Αν δείτε το προφίλ αυτών των ροών είναι πολλωμένο εντελώς. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου μετανάστευση στο μέσο. Υπάρχει πολύ στα χαμηλά εισοδήματα και ελάχιστη στην κορυφή. Οπότε ο καλύτερος τρόπος να το δούμε είναι να δούμε την εξέλιξη αυτών των ε, ομάδων μέσα στον χρόνο. Και έτσι έχουμε μια προοπτική, δηλαδή δεν έχουμε μια στιγμιαία εικόνα όπως είναι το τζίνι, αλλά μας δίνει θα έλεγα μια ταινία αντί για μια φωτογραφία, το, τι, το πώς κινούνται στο χρόνο δηλαδή ο υπομάδες και οι οικογένειες. Αυτό κάνει ο Πάτναμ στις ε, ΗΠΑ και παρακολουθεί την τροχιά ανθρώπων και είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν μιλάμε για τον ρόλο της ευκαιρίας ε, κοινωνικών πολιτικών αναδιανομής. Να δούμε δηλαδή το διαφορετική κατάσταση διαφορετικών ομάδων στην ίδια κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι παρεμβάσεις. Απλά δυστυχώς πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το ρολόι. Έρχομαι λοιπόν στο πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων και θα παρακαλέσω θερμά οι ερωτήσεις να περιοριστούν στο ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς εγγεγραμμένους ομιλητές. Το ίδιο θα περικόψω και τις απαντήσεις Αντί για 10, 7 λεπτά για τους ομιλητές μας. Άρα, 2 με 2,5 λεπτά ο καθένας για τις απαντήσεις τους. Η Ρωμάνα Τόμς, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο εκ μέρους του κυρίου Κάζα, του συντονιστή μας. Λίγα σχόλια και λίγες ερωτήσεις. Φαίνεται να υπάρχει συνένεση ως προς το ότι οικονομικές ανισότητες είναι επιβλαβής για τις κοινωνίες. Υπονομεύουν την ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική σταθερότητα και την πολιτική σταθερότητα. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες κοινωνικές προκλήσεις. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε, τουλάχιστον να μειώσουμε ε, τις ρίζες, τα αίτια των ανισοτήτων θεωρεί επιτακτική πολιτική ανάγκη μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη για την Ευρώπη και επεξεργασία ε, μέτρων για να έχουμε ένα κοινωνικό ευρωπαϊκό τριπλό α στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένε προκλήσει. Ε, οι οικογένειε με χαμηλό εισόδημα πολλαπλασιάζονται και οι διάφορε μελέτε καταδεικνύουν πω όταν η φτώχεια φτάσει και τη μεσαία τάξη αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανάπτυξη και να αποδυναμώσει την κοινωνική συνοχή περιορίζοντα τι ευκαιρίε, όχι μόνο για του ε, λιγότερο ευνοημένου ε, τομεί, αλλά και για όσου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και μια εξωπρεπή διαβίωση να ολοκληρώσω, θα έλεγα, με ρητορικέ κατ' ουσίαν ερωτήσει. Πώ μπορούμε κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο να κάνουμε περισσότερα για του πολίτε μα, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τελικά την αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων με τον σωστό τρόπο. Μήπω θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήσασταν και καλό παράδειγμα προ τη χρήση του χρόνου αγόρευση. Ε, Υπερβάσου Μπερέ από του Σοσιαλιστέ Δημοκράτε για την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ και εγώ το χρόνο αγόρευσης, αλλά το ότι έχουμε δύο επίτροπε σε αυτή την κοινή ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να το τονίσω. Και στρέφομαι και στην επόμενη φάση που είναι αυτή της διατύπωσης προτάσεων. Για τον πρώτο ομιλητή έχω μια ερώτηση. Η σπονδυλική στήλη των ειδικών αναχώρα συστάσεων μήπως θα έπρεπε να είναι αν θέλουμε να έχουμε διόρθωση κατάστασης η εφαρμογή της εγγύησης για την νεολαία. Να είναι αυτή δηλαδή η σπονδυλική στήλη των μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. Για τη δεύτερη ομιλήτρια. Έχω μια ερώτηση για τα φορολογικά, διότι είναι μία από τις πτυχές η οποία αναφέρθηκε. Κατά την άποψή σας λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικότερο μέτρο και έχει γίνει προσπάθεια ορισμένος ε, ευρωπαϊκού δικού χάρτη ώστε τα ευρωπαϊκά φορολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας να προσαρμοστούν καλύτερα στην καταπολέμηση των ισοτήτων. Για τον τρίτο ομιλητή, αφού τον ευχαριστήσω που επέμεινε στην πραγματικότητα αυτή με τους μετανάστες, έναν πληθυσμό πολύ ευνοημένο ή το αντίθετο εντελώς σε πλήρη ένδια. Αυτή η σύσταση Πώ υλοποιείται, ιδίω από του Υπουργού Οικονομικών, δεν θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη στην οικονομική στρατηγική που προτείνεται με αλφαγιώτα. Δηλαδή, οι συστάσει αναχώρα, οι συγκεκριμένε, θα έπρεπε να ευνοούν την υποστήριξη των μεταναστών, την πλαισίωσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή για τον πρώτο γύρο από την Επιτροπή Απασχόληση και από την Επιτροπή, από, συγγνώμη, από την Ομάδα των Κρατών, ο Χάβι Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές μας. Ήταν καταπληκτικέ οι παρουσιάσει τους. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Πρώτον, μιλήσατε κυρίω για τις εισοδηματικέ ανισότητε και αναφερθήκατε στο πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις ανισότητες ε, στον κόσμο και μεταξύ των χωρών. Εγώ όμως θα ήθελα να εστιάσω στις ανισότητες εντός των χωρών της Ένωσης και στην Ευρωζώνη, γιατί τα τελευταία χρόνια οι αποκλήσεις μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης είναι και ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Όταν συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά... Ε, ήταν μια ιδέα και ένα οικοδόμημα που θα αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα και θα δημιουργούσε σε μεγαλύτερη συνοχή και σύγκληση, όχι απόκληση. Το ερώτημα, τι κάνουμε τώρα και πώς επηρεάζουν οι ανισότητες, ιδίως για την Ευρωζώνη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 5-6-7 χρόνια αυτή τη μεγάλη, τη βαθιά ύφεση ε, η πολιτική ε, φορολόγηση, η δημοσιονομική πολιτική, ιδίως για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, ε, το θεματολόγιο τη εσωτερική μεταρρυθμίση, ιδίω στην αγορά εργασίας, ευελιξία κτλ. και η πολιτική των μισθών που πίεσε προς τα κάτω ε, τους μισθούς σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες χώρες γιατί δεν μπορούσε να γίνει νομισματική υποτίμηση άρα θα έπρεπε να υπάρξει νομισμα... Ε, συγγνώμη, μισθολογική υποτίμηση Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι από ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής πλευράς είναι άκρος επιβλαβής αυτές οι ανισότητες ε, και πέραν του αντικτύπου υπάρχει και αντίκτυπος στην υγεία, υπάρχει και αντίκτυπο θεσμικός. Δηλαδή, λόγω των ανισοτήτων, οι κοινωνίες ε, δεν θεωρούνται ότι μπορούν να εκπροσωπηθούν από τους θεσμούς. Και τέλος, υπάρχει και εκλογικός αντίκτυπος και τον βλέπουμε. Πάμε πίσω στους ομιλητές τώρα. Ακολουθώ διαφορετική σειρά, αν το επιτρέπετε. Ο κύριος Ντεβός είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο ακριβέστερα γίνεται, συνδέοντας το θέμα με τη μετανάστευση, με το πρώτο ερώτημα, πώς να επενδύσουμε. Σίγουρα, και συνέγραψα βιβλίο από αυτού, σίγουρα πολλά είδη ε, πράγματα πηγαίνουν στραβά στις αρχές της ε, ηλικίας, στην πρώιμη ηλικία κάποιου. Στο ψηφιακό κόσμο βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει πόλωση, υπάρχει διαφορά στο περιβάλλον, ε, εκπαίδευση κλπ. κλπ. Από όταν είναι καλής, πολύ νέος αρχίζουν αυτές οι αλλαγές. Και η βασική πρόκληση για όλα τα κράτη προνοίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι να αντλήσουν τις πηγές τους, να χρησιμοποιήσουν σε πρώιμο στάδιο της ζωής των πολιτών αυτό που κάναμε σε πιο ομογενή κοινωνία παλιά, που είχαμε κοινή πρόοδο, φυσική κοινή πρόοδο. Η πρόσβαση στην παιδεία παλιά ήταν βασικό εργαλείο που έδινε ίσες ευκαιρίες όλους. Αυτό δεν ισχύει πια. Αυτό πρέπει να επαναξεταστεί. Η οικογενειακή πολιτική ούτως υπήν εν τη ευρία ενία του όρου είναι σημαντικότατο για τους μετανάστες Πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ αφιχθέντων και μεταναστών δεύτερης τρίτη γενιά. Είναι βασικό. Σχεδόν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε και όχι μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγάλο πρόβλημα ενσωμάτωση κάποιων ομάδων μεταναστών που προέρχονται από χώρε εκτό Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάποια χώρα που να πηγαίνει καλά εκεί. Μπορεί να προσπαθήσει κανείς να μάθει τους καλύτερους, αν διερωτηθεί τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, να συντονίσει καλύτερα τη μεταναστευτική ροή μέσω κριτηρίων, μέσω γεωγραφικής κατανομής των μεταναστών. Ανέφερα τις Βρυξέλλες. Ο νεαφιχθής στην Ευρώπη και φτάνει στις Βρυξέλλες. Σκέψου τι τον περιμένει αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια πόλη η οποία είναι πλήρης από μετανάστες σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες τονίες της πόλης. Δεν υπάρχει αξιοπρεπή στέγαση ούτε αξιοπρεπή παιδεία. Ο χειρότερος τόπος να συγγενήσει κανείς ως να είναι εδώ, σε αυτή την πόλη, λόγω ελλείψεως συντονισμού σαν μαγνήτης προσελκύονται όλοι εδώ, διότι εδώ υπάρχει η δικτύωση. Εδώ υπάρχουν άλλοι μετανάστες από την ίδια χώρα που έφτασαν. Οπότε φυσικά κάποιο έρχεται στην ίδια πόλη και πριν το ξέρει κανείς είναι ήδη στο περιθώριο τη κοινωνίας. Η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει κάτι πάνω σε αυτό, ανάντι όσον αφορά την μετανάστευση παρά ε, Όσον αφορά το ευρώ, αν είχαμε θεσμικό βασικό μηχανισμό που απαιτείται για ένα σταθερό ενιαίο νόμισμα, κοινό νόμισμα, δεν θα είμαστε στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, πώς να το πω, τα ημίμετρα, λύσεις μέσω ημιμέτρων. Θα είχαμε μείωση του χρέους και συστημικές α, μεταφορές πόρων στις χώρες νομισματικής ένωσης. Δεν έχουμε φεύγει ακόμα τους κατάλληλους μηχανισμούς ε, πειραματιζόμαστε. Είχαμε αιώνια υποτίμηση, διαθωτικές αλλαγές και όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και αν κολλήσει, κανείς κόλλησε. Αν μπει σε κύκλο κανείς, και επιβάλλει λιτότητα, και η λιτότητα είναι μια λέξη που μπορεί να τη χειραγωγήσει κανείς. Εάν είσαι αυστηρός όσον αφορά τον προπολογισμό και δεν έχεις νέα οικονομική ανάπτυξη φυσική λόγω ελλείψης ζητήσεως και επενδύσεων, κόλλησες. Εμείς θέμε. Είναι πολιτικό σφάλμα, δεν είναι οικονομικό σφάλμα. Είναι θεσμική ευθύνη και νομίζω ότι την Ευρώπη εξαρτάται να λάβει την κατάλληλη απόφαση. Μιλούσαμε για τους νέους και βέβαια είναι τα πρώτα θύματα είναι. Πρέπει να σας διακόψω, λέει ο Πρόεδρος, ήδη χρησιμοποίησατε τα δύο τρίτα του χρόνου των αγορητών. Καταχράστε του χρόνου των άλλων δύο. Συγγνώμη παρεμβαίνω, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Πίκετ έχει το λόγο. Δεν είμαι οικονομολόγος. Οι γνώσεις μου αφορούν την υγεία του πληθυσμού και κατανόηση κοινωνικών, οικονομικών δικτών που καθορίζουν την υγεία των πολιτών. Θα αφήσω παράμερα το ερώτημα ποια κατεπήγοντα φορολογικά μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στου εμπειρογνώμου θα αφήνω αυτό. Υπάρχει ένα έγγραφο με τίτλο Έκκληση για αλλαγή ε, από το Επιστημονικό Συμβούλιο η Προοδευτική Οικονομία εκδόθηκε, το στηρίζουν στους δημοκράτε τη Ευρωπαϊκή συνεγράφει από τον Τζον Στίγκλε, τον Ζαν Πολ Φιτούση και πολλού άλλου οικονομολόγους... και από την υποφαινομένη. Να πω κάτι όσον αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία που έχουν οι διαφορέ στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Δηλαδή, πώ η λιτότητα, το πώ επευλήθη η λιτότητα σε κάποιου πληθυσμού. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα σε μια συνεδρίαση στη Βαρκελόνη του Διεθνού Δικτύου για την έρευνα για ανισότητες στην παιδική υγεία και αρχίζουμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο που έχει η λιτότητα στην υγεία των παιδιών στις χώρες εκείνες στις οποίες έχει επιβληθεί η λιτότητα. Πέρασε κάποιος χρόνος να δούμε την επιρροή στα στοιχεία, αλλά βλέπουμε αλλαγές όσον αυτά τα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών, την σημότητα βρεφών στα επίπεδα του στρες, διατροφικό καθεστώς κλπ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τους πρώτες ενδείξεις μιας αυξήσεως νησιμότητας μεταξύ των πλέον ηλικιωμένων μετά τη λιτότητα. Είναι η πρώτη φορά που η θνησιμότητα στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε και δεν μειώθηκε από όταν άρχισαν μετρήσει. Και εμεί ξεκινήσαμε τι μετρήσει από πολύ παλιά, πριν από του άλλου. Έχουμε πάνω από έναν αιώνα μειώσει θνησιμότητα και τώρα βλέπουμε αύξηση τη θνησιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο, ο κ. Πίρσον, ο ο σημαντικό ομιλητή, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολύ σύντομα. Καταρχά, ετέθη ένα ερώτημα για, το μέσο, για την εγγύηση για την νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικότατο αυτό θέμα. Δείχνει η δουλειά μα ότι αν δεν καθιερωθεί στην αγορά εργασία, αν δεν δημιουργήσει καριέρα την πρώτη δεκαετία μετά την είσοδο στην αγορά εργασία, ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί μετά στην οικονομία, ποτέ δεν θα καλύψει το κενό. Υπάρχει μια χρονική περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Το βλέπει αυτή κανείς βλέποντας τι έγινε, πηγαίνοντας πίσω πριν από 40-50 χρόνια. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν καθιερωθεί τότε, ποτέ δεν κατάφεραν να καλύψουν την υστέρηση. Πρέπει η νεολαία να ξεκινάει από καλή βάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν λεπτομέρειε όσον αφορά την εγγύηση για την νεολαία κλπ. Πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά η κεντρική ιδέα είναι σωστή. Δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να επανέλθω είναι η άλλη ιδέα του αντικτύπου που έχει η μετανάστευση στι ανισότητε. Υπάρχει ένα αντίκτυπο, αλλά λυθεύει επίση ότι όσο καλύτεροι είμαστε στην ένταξη των μεταναστών, τόσο μικρότερο ο αντίκτυπο. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξο από πολλού άλλου. Δηλαδή, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την ένταξη, κυρίω σε κάποιε χώρε ε, στην Ευρώπη, είναι ότι τα κάνουμε όλα λάθο. Το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει οι πρόσφυγε μετανάστευση να πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν δουλειέ και όχι εκεί που είναι η στέγαση, όχι εκεί που είναι τα σχολεία, όχι εκεί που βρίσκεται το σύστημα υγεία. Πρέπει να πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν δουλειέ και να εξασφαλίζεις ότι ο κόσμος θα βγαίνει από ειδικά σχήματα ε, εκπαιδευτικά ή απασχόληση στο ταχύτερο δυνατόν. Αν μιλά για πρόσφυγε, να εξασφαλίσει ότι οι πρόσφυγε θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία στο ταχύτερο δυνατόν. Αυτό δεν βασίζεται επί κάποια ε, προκατάληψης, αλλά σε αρκετά στοιχεία που έχουμε συλλέξει από διάφορες χώρες για την επιτυχία που έχουν διάφορες ομάδες όσον αφορά την ένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα απεσιόδοξοι. Είναι ένα πρόβλημα σίγουρα, αλλά μπορεί να το λύσουμε. Τρίτο σημείο τελικά που θέλω να αναφέρω, ναι συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να επενδύσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην παιδεία των νέων παιδιών, ακόμα και πριν την γέννηση, άμα πάμε, αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια τάση από πλευρά των πολιτικών να προσπαθούν να βρουν την μαγική λύση για την εξίσωση των ευκαιριών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν υπάρχει κάποιο τρόπο εξισώσεω των ευκαιριών που δίνονται στι κοινωνίε, αν δεν εξισώσουν επίση και τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να βρει πολιτικέ οι οποίε εξισορροπούν μεγάλε ανισορροπίε μεταξύ των συνδυμάτων των γονέων. Μόνο αντιμετωπίζοντα τα αποτελέσματα καθώ και τι ευκαιρίε, μπορείς να περιμένεις να έχεις καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά και αυτό τότε μας οδηγεί σε μελλοντική ανάπτυξη. Αυτά και ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο, την κυρία ούφσκοκ την εκπρόσωπο της Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. θα δώσω το λόγο στον κύριο Λούνς που εκπροσωπεί το ECR στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο μου προξενεί εντύπωση στη συζήτηση αυτή είναι ότι έχει αλλάξει η εστίαση της συζήτησης. Δεν μιλάμε πλέον για ατομική ευθύνη, αλλά μιλάμε για εξωτερικούς παράγοντες. Όταν είναι επιχειρηματίας επιτυχής, δεν είναι κάτι το οποίο έκανε ο ίδιος, αλλά ήταν τυχερός. Όταν έχει κάποιος δυσκολίες, είναι θύμα, είναι άτυχος. Και το ακούω και σήμερα, κυρίως αυτά τα οποία είπε η κυρία Πίκετ, είστε επιτυχημένη επιδημιολόγος. Έχω την εντύπωση πως ε, δεν ξέρω ε, εάν θα αντιμετωπίζατε μια πανδημία με τον ίδιο τρόπο, με μια αναδιανομή των εμβολίων και θα πηγαίναν όλα καλά. Κοιτάξτε, ε, βλέπετε νομίζω την ανισότητα ως μια αρρώστια, ενώ έχει θετικές πτυχές. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των ίσων ευκαιριών οπωσδήποτε, αλλά αντιλαμβάνομαι και τους κινδύνους της μεγάλης και κεντρικής αναδιανομής. Και πραγματικά δεν βλέπετε κι εσείς αυτή την ε, διαφορά. Παραδείγματος χάρη βλέπετε το τι γίνεται στην Ελλάδα, όπου πηγαίνουμε και σε λιγότερη ανάπτυξη και θα έχουμε και δυσκολότερες καταστάσεις ε, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα με την εστίαση στην αναδιανομή. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ρόμπερτ Τσίλ που εκπροσωπεί την ομάδα του ECR επίσης ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ γιατί είχα να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία. Εγώ ζούσα σε μια ίση ε, χώρα, τη Σοβιετική Ένωση ε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχε ακριβώς, ε, δεν δημιουργούσε και μια ευχάριστη κατάσταση η ευτυχία και τώρα είναι πολύ πιο άνηση βεβαίως η Λετωνία αλλά τελείως διαφορετική κατάσταση. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν Είπατε πως δεν υπάρχει αναδιανομή μέσω του συστήματος ε, επιδομάτων κλπ. Γιατί, γιατί όλες οι κυβερνήσεις αριστερά ή δεξιά είναι υπέρ της, κοινωνική της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Επίσης ε, λέτε πως η αναδιανομή, η ασθενέστερη ε, δεν σημαίνει ότι έχει σχέση με το αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Καμιά φορά οι οικονομολόγοι μιλάνε και λένε ότι η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος είναι σημαντική για τις επενδύσεις. Συμφωνείτε. Για του άλλου ομιλητέ, επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε κάποια σχόλια για ένα συνολικό, για ένα ε, εισόδημα κοινό το οποίο προσφάτως καταψηφίστηκε στην Ελβετία. Θεωρείται ότι είναι κάποια μαγική λύση. Και η άλλη ερώτηση αφορά το κοινωνικό dumping. Εδώ πέρα παλεύουμε θα έλεγα με το κοινωνικό ντάμπινγκ σε πολλούς τομείς στην ενιαία αγορά, στις μεταφορές και αλλού θεωρείται πως ε, αν το αντιμετωπίσουμε θα υπάρχει περισσότερη ισότητα στο επίπεδο της Ένωσης ή το αντίθετο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, then I'll give the floor. Ευχαριστώ. Πρόσωπος της Άλμπε, παρακαλώ, και για τις δύο επιτροπές, Έμπλ και Έκον. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτά τα τρία λεπτά και πρώτον θα κάνω κάποιες οικονομικές παρατηρήσεις ως εκπρόσωπος Επιτροπής ΕΚΟΝ στη συνέχεια. Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω όντας συναισθηματικά φορτισμένος και να ευχαριστήσω καταρχάς τους προσκεκλισμένους μας που μας δώσανε πολύ θετικέ πληροφορίες αλλά ως εισηγητής της έκθεσης κατά της ανισότητας θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, πιο άμεσος και να ανταποκριθώ περισσότερο στη συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει μια δυναμική ανισότητα σε αυτή τη στιγμή στις κοινωνίες μας, καθώς προσπαθούμε να βγούμε από την κρίση. Από οικονομικής λοιπόν πλευράς πιστεύω ότι η διόρθρωση της δυναμικής αυτής ανισότητας θα έρθει από την οικονομική πολιτική και όχι από τις κοινωνικές πολιτικές που θα μας απασχολήσουν στο δεύτερο τμήμα της παρέμβασής μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο δυναμικής ανισότητος που ζημιώνει αυτή τη στιγμή την ίδια την ανάπτυξή μας, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερη ανεργία και περισσότερη ανισότητα κατά, την, κατά συνέπεια. Συνεπώς, έχω να κάνω την εξή ερώτηση. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν θα πρέπει να παρακολουθούμε και τη δυναμική της ανισότητας. Έχουμε το συντελεστή Τζίνι, ο οποίος μπορεί να μην είναι τέλειος, Υπάρχουν και άλλοι στερεστέ πάλμα, για παράδειγμα, που ενδεχομένω να είναι καλύτεροι. Για ποιο λόγο να μην παρακολουθούμε μέσω των στερεστών αυτών την ανισότητα και να κάνουμε συστάσει για την δημοσιονομική πολιτική, για την πολιτική επενδύσεων, για την παιδεία, συστάσεις ε, όσον αφορά τις τομεακές πολιτικές, όπως η επιλογή των τομέων επί των οποίων θα πρέπει να επέμβουμε και ούτω καθεξής. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τα βαθύτερα αίτια της ανισότητος. Όσον αφορά τώρα τις κοινωνικές πτυχές, τα κοινωνικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται θεωρώ ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν διορθωτικά. Έρχονται απλώς να απαλύνουν κάποια προβλήματα. Σαφώς είναι απαραίτητα τα κοινωνικά αυτά μέτρα, λειτουργούν ανακοφιστικά, σαφώς θα πρέπει οι πολίτες μας να υποφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά α μην θεωρούμε ότι τα κοινωνικά αυτά μέτρα είναι μέτρα διόρθωση. Στα πλαίσια λοιπόν των κοινωνικών πολιτικών έχουμε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή. Σαφώ θα πρέπει να έχουμε τέτοια κοινωνικά μέτρα, που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κιόλα. Και επανέρχομαι στην οικονομική πτυχή. Στόχο τη οικονομική μα πολιτική θα πρέπει να είναι η ικανότητά μα να χρηματοδοτούμε τι κοινωνικέ πολιτικέ, προκειμένου να έχουμε πιο συνεκτικέ κοινωνίε. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προπόθεση τη μετέπειτα μάχη που θα πρέπει να δώσουμε κατά τη ανισότητα. Ευχαριστώ. Thank you. I will now give the floor to Madam... Ευχαριστούμε. Η κυρία έχει Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να, με, να μετρήσει κανείς την ανισότητα που επικρατεί στην Ευρώπη. Κάποιοι όμως έχουμε το θλιβερό προνόμιο να επιβεώσουμε ως στατιστικές και με τα ίδια μας τα μάτια. Ως Ευρωβουλευτής κινούμε ανάμεσα σε μια από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης που είναι το Βέλγιο, στην πιο φτωχή που είναι η Βουλγαρία όπου γεννήθηκα και σε αυτή που έχει χτυπηθεί πιο πολύ από την κρίση και τη λιτότητα την Ελλάδα όπου έχω εκλεγεί ως Ευρωβουλευτής. Φυσικά όταν μιλάμε ανισότητες οι διαφορές είναι δραματικές. Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν τη χαμηλότερη αμοιβή εργατόρες ως και 2 ευρώ, όταν στη Δανία είναι 35 ευρώ και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει σχεδόν 20 ευρώ. Ο κατατάτος μισθός στη Βουλγαρία είναι 180 ευρώ, όταν στο Λουξεμβούργο φτάνει το 1900 και στο Βέλγιο 1500 ευρώ. Γιατί όμως, γιατί η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό του ανήλικου πληθυσμού, το 40% σε κίνδυνο φτώχειας, όταν τη Τσεχία είναι 15% και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 11%. Γιατί η Ελλάδα έχει πενταπλάσιο ποσοστό ανεργίας από την Γερμανία, γιατί ο κατώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 20 φορές πάνω από το κατώτατο μισθό στη Βουλγαρία, γιατί η Ελλάδα έχει έναν από τους χειρότερους δείκτες γονιμότητας. Μόλις 1,30 ο αριθμός παιδιών που αντιστοιχεί ανά γυναίκα σε ηλικία αναπαραγωγής σε σύγκριση με χώρες που έχουν μικρότερο πληθυσμό, όπως Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, με καλύτερο δίκτυο γονιμότητας. Γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια τάση αυτά τα φαινόμενα ανισότητας να τα αντιμετωπίζουμε ως αποτυχία της κάθε χώρας και της κοινωνίας της να αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια ως αποτυχία του ίδιου του φτωχού ή την ανεργία ως προσωπική αδυναμία του ανέργου. Αυτές τις απόψεις τις κάνουμε μερικές φορές ακόμη και από εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας. Λέγεται συχνά από την Κομισιόν ότι για την κατάσταση της φτώχεια ή της υψηλής ανεργίας σε ορισμένες χώρες φταίει το ότι δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις είναι ένας πολύ επικίνδυνος μύθος που δίνει τροφή σε εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις. Το βλέπουμε τώρα στην περίπτωση της Βρετανίας. Η εκστρατεία υπέρ του Brexit στηρίζει στον μύθο ότι πρέπει να σταματήσει η Βρετανία και ο Ευρωπαϊκός Βορράς να πληρώνει τους τεμπέλεδες του Νότου. Η αλήθεια είναι ότι η ανισότητα δεν είναι αποτυχία των φτωχότερων, αλλά αποτυχία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί για σύγκληση, έχουμε απόκληση και αύξηση των ανισοτήτων. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ελλάδα, που μέσα από έξι χρόνια στο μνημόνιο χειροτέρεψε η κατάσταση της σε όλους τους δείκτες της ανισότητας και της στόχιας. Γιατί συμβαίνει αυτό η ευρωπαϊκή οικονομία ω σύνολο λειτουργεί ω μηχανισμό μεταφορά μεταφοράς πλούτου από την περιφέρεια στο κέντρο, από το φτωχότερο νότο στο πλουσιότερο βορρά, μέσα από τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα 5-6 χωρών. Αυτή είναι η κυριότερη ανισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κανείς δεν τολμάει να αντιμετωπίζει ένα μη τυγείο εθνικός εγωισμός των ισχυρότερων και πλουσιότερων χωρών. Και όμω, αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισορροπία σε λίγα χρόνια, όχι μόνο τα μετράμε ακόμη πιο εκρηκτικές ανισότητε, αλλά τα είναι αδύνατο να κρατήσουμε μια ελάχιστη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Λυπή, ε, μάλλον θα δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές, ε, κυρία Πικέτ. Λυπούμε και είμαι απογοητευμένη που χρειάζεται να απαντήσω ε, το ερώτημα του πρώτου βουλευτή που μάλλον δεν μας άκουσε πολύ καλά. Εγώ δεν ζήτησα να υπάρχει αναδιανομή μόνο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Είπα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι, μεγαλύτερη οικονομική δημοκρατία και ε, η μείωση των προφόρων, αλλά και οι τρεις μας νομίζω είπαμε ότι βάσει των αποδείξεων που έχουμε και των εμπειριών μας και τα λοιπά, θεωρούμε ότι με την ανισότητα μειώνεται η οικονομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ε, κίνδυνος προς την οικονομία, ε, δηλαδή με το να κάνουμε κάτι για τις ανισότητες. Το αντίθετο, αν δεν κάνουμε κάτι έχουμε κίνδυνο για την οικονομία. Και νομίζω ήταν σαφές και, για... και το είπαμε και τρεις και λυπούμε που πρέπει να επαναλάβω κάτι που το είπαμε και τρεις. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω ε, στον κύριο που μίλησε για την υγεία. Φυσικά και υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που οδηγούν σε δυσαρέες και σε προβληματίες και τα λοιπά. Ε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι απλά μια συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι με τις ανισότητες μειώνονται οι οι καλές συνθήκες ε, και είδαμε να μειώνεται και το προσδόκιμο ζωής στις χώρες που μελετήσαμε στη δική μας έρευνα, κυρίως αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση ανισοτήτων με βάση τα στοιχεία ε, στο British Medical Journal εδώ και χρόνια. Επίσης, συζητούμε συνεχώς για, τη, ε, για την παιδεία. Έχω να τονίσω το εξή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι δάσκαλοι και τα σχολεία να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι ανισότητες για τη ζωή ζωή των γονιών και των οικογένειών Βλέπουμε ψυχική υγεία σε, ανισο... σε κοινότητε με Βλέπουμε ψηλά επίπεδα εθισμών, ε, διασπάσει οικογενειών, ε, προσωπικά ε, χρέη, πάρα πολλέ ώρε εργασία κτλ. Πώ μπορεί κανεί να περιμένει υπό τέτοιε συνθήκε τα σχολεία να φτιάξουν, να διορθώσουν τη ζημιά τη ανισότητα είναι ε, σαν να προσπαθούμε να σφουγγαρίζουμε ε, χωρίς να έχουμε κλείσει τη βρύση όμως. Ε, πώς θα λύσουμε έτσι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κύριο Πίρσον. Ναι, ευχαριστώ. Να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη αναδιανομή όπως παλιότερα. τονίζω, δεν μιλάμε εδώ για ποσά φόρων και εμβασμάτων στην οικονομία, αλλά το ποσοστό της αναδιανομής ανακατανομής αυτών των ποσών. Και πραγματικά παρατηρούμε πτώση, σημαντική πτώση. Βέβαια ε, υπάρχουν κάποιες καμπανεβάσματα ανάλογα με τον πολιτικό κύκλο, αλλά η μακροχρόνια τάση είναι λιγότερο αναδιανεμητική φόρη και ε, ε μεταφορές. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπήρξε μείωση των δαπανών και κοινωνικών επιδομάτων ε, στις διάφορες οικονομίες για να δοθούν περισσότερα κίνητρα για εργασία. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό. Τι δεν έγινε όμως, οι συντάξεις ε, δεν τις ακούμπησαν, τις παλιότερες, τις μελλοντικές ναι, όχι όμως τις σημερινές. Η σύνταξη δηλαδή βασίζεται στις προηγούμενες εισφορές και είναι το λιγότερο αναδιανεμητικό τμήμα του συστήματος ε, φόρων και επιδομάτων συνήθως. Βλέπουμε όλο και λιγότερη αναδιανομή. Τώρα, το δεύτερο, φορολογία. Στην Ευρώπη και αλλού έγινε εστίαση κυρίως στους φορολογικούς συντελεστές και όχι στη φορολογική βάση. Στην πιο ακραία περίπτωση βέβαια, και γι' αυτό και έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση, φορολογικούς παραδείσους, φορο κτλ. Αλλά είναι ευρύτερο το πρόβλημα, ακόμη και όταν έχουμε ε, νόμιμα ε, κάποια μέτρα, δεν νομίζω ότι η νόμιμη φοροαποφυγή ε, αντιμετωπίζεται. Πρέπει να έχουμε την ευρύτερη δυνατή φορολογική βάση. Για αυτούς τους δύο λόγους βλέπουμε ότι η δύναμη του συστήματος προνοίας έχει μειωθεί. Ευχαριστώ, κύριος Δεβός. Ε, ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ντεφός. Ε, δεν θα μιλήσω μόνο εγώ αυτή τη φορά για το πρώτο ερώτημα είναι δύσκολο να προσπαθήσω να το απαντήσω. Μπορούμε να δούμε την ανισότητα με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, διαφορετικές αιτίε, συνέπειες. Εγώ θα αναφερθώ στο έργο του Μπρανκο Μιλάνοβιτ, ε, οικονομολόγου της Παγκόσμια Τράπεζας, που είπε ε, ότι είναι σαν την χολυστερίνη. Υπάρχει καλή και κακή χολυστερίνη και πρέπει να γίνεται η διάκριση από πλευρά ε, πολιτική. Τώρα, θα ήθελα να αντιδράσω σύντομα στο ερώτημα για ένα ε, γενικό βασικό εισόδημα, ευρύτατο ζήτημα, αλλά καθαρά από τη σκοπιά της ανισότητας ε, νομίζω πως ε, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει περισσότερη ανισότητα και να εδρεώσει την ανισότητα. Είναι ένα μέτρο με το οποίο αισθανόμαστε καλά αλλά για αυτούς οι οποίοι θα το λαμβάνουν θα έχει πιθανώς ε, καταστροφικά αποτελέσματα. Το θέμα του κοινωνικού dumping. Πάλι εδώ πέρα ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου. Αν είναι dumping, είναι dumping και δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή η λέξη dumping ε, υπονοεί μια παράνομη πρακτική. Αλλά η απόσπαση, αυτό το οποίο λέτε δηλαδή, κάποιο ο οποίο είναι στην αγορά εργασίας μια χώρα και πάει προσωρινά σε μια άλλη, μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη, για να αναφερθώ και στη Βουλγαρία, θα προχωρήσει σε μια σύγκληση μεταξύ ευημερία και ε, δουλειών στην... μεταξύ κρατών μελών. Το πρόβλημα είναι βεβαίω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει χειραγώγηση του συστήματος και βεβαίω δεν υπάρχει ανάληψη της ευθύνης, ε, δεν υπάρχει μια συνοχή στην πολιτική μεταξύ των κρατών μελών που στέλνουν και εκείνων που λαμβάνουν τα άτομα, τα αποσπασμένα. Γι' αυτό υπάρχει ακριβώς η δυνατότητα κατάχρησης ε, του συστήματος. Είναι πιο πολύ πολιτικό παρακονομικό ζήτημα. Και σταματάω. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον Μάρκο Τσάνι, 1,5 λεπτό. Εγώ θα μιλήσω και για τις δύο επιτροπές, οπότε πρέπει να έχω τρία λεπτά. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερις γρήγορες ερωτήσεις για τους ομιλητές μας. Πρώτον, όσον αφορά τα βαθύτερα αίτια της ανισότητας θεωρώ ότι ε, ο γενικότερος και πιο σημαντικός λόγος είναι το αναπτυξιακό κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο το οποίο έχουμε σήμερα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το μοντέλο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Ποιε είναι οι επιπτώσει ενός τέτοιου κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου όσον αφορά την ανισότητα βασιζόμενη στις καταπληκτικές έρευνες του κυρίου Στίγκλιτς. Δεύτερη τώρα ερώτηση. Αυτή αφορά την Ευρωζώνη και το ανέφερε συνάδελφος από τους αριστές πριν από λίγο. Το μοντέλο αυτό οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται προφανώς με το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Είδαμε όμως ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί τεράστια ανισότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χώρες δανειστές και χώρες οι οποίες δανείζονται. Έχουμε χώρες οι οποίες μπορούν αυτή τη στιγμή να λειτουργούν με συναλλαγματική ισοτιμία πολύ ψηλή και άλλοι με ισοτιμία πολύ χαμηλή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό με τη σειρά του έχει επιπτώσει στους ίδιους τους πολίτες και έχει επιπτώσεις και στις πολιτικές που τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν να προωθήσουν ή θα μπορούσαν να προωθήσουν για να μειώσουν τα φαινόμενα ανισότητας. Ας μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα μόνιμων μεταφορών πόρων όπου οι πιο πλεονεκτούσες χώρες θα κληθούν τελικά να βοηθήσουν τις ε, χώρες που το έχουν μεγαλύτερη ε, ε, ανάγκη. Αυτό το είχαμε δει στο παρελθόν και στην Γερμανία όπου υπάρχουν πολλά λάντερ, πολλά κρατήδια της Γερμανίας τα οποία ζουν μόνο και μόνο επειδή ακριβώς υπάρχει μεταφορά πόρων και χρημάτων από κρατήδια της Γερμανίας, κυρίως στη Δυτική Γερμανία. Ο εκπρόσωπος του ΟΣΑ μίλησε για μία ανισότητα η οποία αυτή τη στιγμή είναι βαθιά ριζωμένη. Έχει όμως μια γενεαλογική πτυχή η ανισότητα αυτή. Μπορούμε να πούμε ότι από τη μία γενιά στην άλλη τα φαινόμενα ανισότητας μπορεί να μειωθούν η δικιά μου γενιά, που είναι η γενιά των millennials στις δεκαετίες του 2000, είναι μάλλον η πρώτη γενιά μετά τον πόλεμο, η οποία αντιμετωπίζει περισσότερες πλέον δυσκολίες από ό,τι οι πατέρες και οι μητέρες μας, η προηγούμενη δηλαδή γενιά. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για την διαγενεολογική διάσταση του φαινομένου της ανισότητας. Οι πολιτικές που προσπαθούμε να υιοθετήσουμε αυτή τη στιγμή κάνουν κάτι για το ζήτημα αυτό. Τα όσα γίνονται στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Γαλλία έχουν ως στόχο να μειώσουν τις ανισότητες από τη μία γενιά στην άλλη. Ευχαριστούμε. Γιάν Κέλλερ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις για τον κύριο Μαρκ Πίρσον. Πρώτον, Αναφερθήκατε σε μια αύξηση της ανισότητας όσον αφορά το εισόδημα. Πολλοί ερευνητές όμως για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μας λένε ότι αυτό το οποίο αυξάνεται ακόμα γρηγορότερα είναι η ανισότητα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Ο Λίσεβέλ στην Γαλλία μιλούσε για το φαινόμενο αυτό και υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο σχετικά με το φαινόμενο αυτό του κληρονομικού καπιταλισμού. Πιστεύετε λοιπόν ότι οι κοινωνίες που έχουν μια τέτοια ανισότητα ως προς την ιδιοκτησία, ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, θα δούνε και μια εισοδηματική ανισότητα στο μέλλον. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε διάφορους λόγους οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανισότητα. Αλλά δεν είπατε τίποτα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις δυστυχώς. Είναι και αυτός ένα σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει από τη δεκαετία του 80 και μετά στα φαινόμενα ανισότητας από τη δεκαετία του 80 και μετά άρχισε να αυξάνεται πολύ περισσότερο και η ίδια ανισότητα. Οι πολυεθνικέ αυτέ επιχειρήσει τοποθετούν θέσει απασχόληση σε χώρε με χαμηλότερη προστιθέμενη αξία και με χαμηλότερε μισθολογικέ απαιτήσει στην Ευρώπη. Ενώ θέσει μεγαλύτερη ευθύνη τι θέτουν σε χώρε με μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. 400 εκατομμύρια κορώνες αυτή τη στιγμή φεύγουν από τη χώρα μου κάθε χρόνο. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ, ένα 10% του ΑΕΠ μας πηγαίνει σε πολυεθνικές επιχειρήσεις σε αιτήσια βάση. Και παράλληλα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η τσεχική δημοκρατία δαπανεί ένα 20% του ΑΕΠ της για κοινωνικά επιδόματα, ενώ μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 28,5% είναι σύμπτωση το ότι οι χώρες της Ευρωζώνης δαπανούν 400 δισεκατομμύρια κορώνες τσεχικές περισσότερο από ό,τι μπορεί ποτέ να δαπανίσει η ίδια η χώρα μου. Ακριβώ επειδή εμεί τα χρήματα αυτά που θα πρέπει να τα δίνουμε σε κοινωνικέ πολιτικέ, τα δίνουμε τελικά σε πολυεθνικέ επιχειρήσει. Πώς μπορεί λοιπόν να μειωθεί η ανισότητα ανάμεσα στις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν μειώσετε όλες αυτές τις εκροές πόρων προς πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αν δεν μείνουν στις χώρες μας τα χρήματα αυτά δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να προωθήσουμε κοινωνικές πολιτικές. Το λόγο τώρα έχει ο τελευταίος ομιλητής, η κυρία Τόμσεν που εκπροσωπεί το ΕΛΚΑ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη φορά θα ήθελα να μιλήσω σλοβενικά, διότι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που αφορά τη χώρα μου, που δείχνει ότι άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη. Ακούσαμε προσεκτικά την παρουσίαση και θα είδατε ότι η Σλοβενία πραγματικά είναι η πρώτη χώρα όσον αφορά τους ε, δείκτες ανισότητας. Και θεωρείται ότι είναι καλό σαν μαντάτο. Γνωρίζοντας τη χώρα μπορώ να πω ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο ρόδινη. Λοιπόν πέρσι είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έφυγαν από τη Σλοβενία, την εγκατέλειψαν, διότι η κατάσταση είναι αφόρητη. Είμαι κατά της ανισότητας του εισοδήματος, ταυτόχρονα όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι και ένα νόμισμα με δύο υπόψεις. Ένα λεπτό θα έχετε. Και αυτό διότι ο συνάδελφος της Επιτροπής Απασχόλησης πήρε χρόνο. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Θα ήθελα να πω ή να ρωτήσω το εξή. Όταν κάνετε τις αναλύσεις σας αυτές, λαμβάνετε υπόψη το λόγο για τον οποίο μόνο τις χώρες, Λουξεμβούργο, Γερμανία και Πολωνία, εποχές κρίσης μπόρεσαν να μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ των φτωχών και εκείνων που είναι πλούσιοι. Κάνατε μια ανάλυση του όλου ιστορικού, τι βήματα έγιναν ούτω ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερες ανισότητες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Βλέποντας τις ανισότητες, κυρίως τις οικονομικές ανισότητες, ποια είναι η μορφή η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τη συγκρίνει κανείς με άλλες υπήρους Υπάρχει λοιπόν κάποια σύγκριση, διαφορά εικόνας μεταξύ Ευρώπης και άλλων υπήρων. Σας ευχαριστώ. Ξεκινήσουμε με τον κύριο Πίρσον. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ε, θα είμαι σύντομος, γιατί ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό των γενναιών. Πράγματι, η αύξηση των ανισοτήτων δεν ε, ε, είναι ίσο κατανεμημένη μεταξύ γενεών. Εάν χωρίσουμε τον πληθυσμό σε γενιές, οι τωρινοί τριαντάριδες είναι πολύ πιο άνηση από την προηγούμενη γενιά όταν ήταν 30 και πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο επαναλαμβάνεται για τα δύο τρίτα των χωρών, όχι παντού. Στις περισσότερες χώρες είναι λοιπόν γενεακή η αύξηση της ε, ανισότητας. Δεν είναι λοιπόν ότι είναι πιο φτωχές οι επόμενες γενιές, αλλά είναι πιο άνισες. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά εντός των γενεών. Δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα του πλούτου. Σωστά, εγώ μίλησα μόνο για το εισόδημα. Τώρα αρχίζουμε να έχουμε δεδομένα για την Ευρώπη, για την ανισότητα του πλούτου και είναι σοκαριστικά όσον αφορά την συγκέντρωση του πλούτου. Ε, δηλαδή το εισόδημα οχριά μπροστά στην ανισότητα του πλούτου. Ε, στο βαθμό που μιλάμε για το 1% της Ευρώπης που έχει ίσως ε, γύρω στο 50% του πλούτου. Όταν λέμε γιατί το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και η Πολωνία μείωσαν την ανισότητα. Κοίτα, βασικά έμεινε σταθερή η ανισότητα και αυτό λόγω της πολύ καλής απασχόλησης, ειδικά σε Γερμανία και Πολωνία, ε, οι γυναίκες οι οποίες μπήκαν στην αγορά εργασίας. Αν δείτε την περίοδο της κρίσης, ναι, Βεβαίω και εκεί ισχύει, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν υπονοούμε ότι η οικονομική κρίση ε, αυξάνει οπωσδήποτε την ανισότητα. Δεν το έκανε στην αρχή, γιατί είχε φάσεις. Στην πρώτη φάση της οικονομικής κρίσης έπεσε η ανισότητα στην Ευρώπη και αυτό κυρίως επειδή ξοδέψαμε περισσότερο σε μέτρα αναζωογόνησης οικονομίας, σε κοινωνικές παροχές και μειώσαμε και τους φόρους σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο αντίκτυπος ήταν να μειωθεί η ανισότητα. Μετά όταν περάσαμε στην λιτότητα βλέπετε μια διεύρυνση της ανισότητας. Οπότε η εξέλιξη της ανισότητας στο χρόνο είναι πολύπλοκη. Νομίζω τελείωσε ο χρόνος μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πίκετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, λίγα πράγματα. Μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία για την ανισότητα του πλούτου, μόλις πρόσφατα μπορέσαμε να δούμε το ζήτημα σε σχέση με την υγεία του πληθυσμού, αλλά η εικόνα είναι η ίδια με το εισόδημα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα του πλούτου, η υγεία είναι χειρότερη. Κοιτώντας την δεκαετία 2000-2009 μπορέσαμε να δείξουμε ότι οι αλλαγές στην ανισότητα του εισοδήματος σχετίζονται με τις αλλαγές στην υγεία των παιδιών. Η Σουηδία που έχει αυξανόμενη ισότητα βλέπουμε ότι έχει μία μείωση της ε, ευημερίας των παιδιών όπως θα περίμενε κανείς. Οπότε αρχίζουμε μία μακρόχρονη ανάλυση που κοιτάει τις αλλαγές στην ισότητα και το τι ε, αντίκτυπο έχουν και ενισχύουν την εικόνα που ανέφερα. Το τελευταίο θέμα για την Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, σε γενικές γραμμές η Ευρώπη είναι μια πολύ πιο ίση ε, περιοχή του κόσμου, αν και υπάρχουν διάφορε, αλλά είναι μια ε, περιοχή η οποία δεν πηγαίνει προς περισσότερη ισότητα, αλλά προς λιγότερη. Η μόνη περιοχή του κόσμου που πηγαίνει σε βελτίωση είναι η Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχουν πολιτικές όπου βασίζεται σε πολιτικές αποφάσεις. Οπότε οι περισσότερες ε, ίσες χώρες είναι στην Ευρώπη, αλλά πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντεφός. Ναι, γρήγορα νομίζω πρέπει να τονίσουμε το ότι πρέπει να περιλάβουμε τον πλούτο, το κεφάλαιο πράγματι. Υπάρχει... Αυτή είναι η προσθέμενη αξία του Τόμας Πικετή η ε, στη συζήτηση τη μεθοδολογία του πώς θα αξιολογήσουμε τον ε, πλούτο δεν είναι εύκολο και το τι συνέπειες έχει η συγκέντρωση του και η συσσόρευση του πλούτου είναι ανοιχτό αυτό προς συζήτηση ε, είναι κάτι το θετικό όμως Είδα να δούμε την φορολογική δικαιοσύνη, είχαμε τρεις γενιές ειρήνης, παγκοσμιοποίηση, μια μετακίνηση προ το χρηματοπιστωτικό τομέα, οπότε λογικό είναι η συγκέντρωση του πλούτου να είναι άνηση και βεβαίω αν δούμε μια συνολική φορολογική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Τονίζουμε εδώ πέρα, εγώ τονίζω την πτυχή των γενεών που θεωρώ ότι λείπει αυτή η συζήτηση και τέλος υπήρχε ένα ζήτημα για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Νομίζω και πάλι ότι δεν είναι οριστική η κρίση αυτού του πράγματος, ε, το τι αποτέλεσμα έχει. Υπάρχουν δύο πτυχές. Η κλασική ρύθμιση της αγοράς εργασίας που θέλει να προστατεύσει τις δουλειές από την οικονομική αλλαγή που έχει οδηγήσει σε κατακαιρματισμό στην αγορά εργασίας ε, μεταξύ των παλαιών και των νέων ε, που δεν μπορούν να προσληφθούν γιατί βεβαίως κοστίζει πάρα πολύ το να προσλάβουμε έναν προστατευμένο υπάλληλο. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι καλό για την ανισότητα. Και αν δούμε την δυναμική ε, της σταδιοδρομίας, την ταινία όπως είπατε για την η φωτογραφία, α, δεν είναι καλό. Ε, το άλλο θέμα είναι να πούμε πώς θα ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό, να μπουν περισσότεροι στο σύστημα. Αυτό θα είναι το ιδανικό μείγμα πολιτικής, αν υπάρξει μια ε, ελαστικοποίηση του καθεστώτος της Ρωσίας. Αυτό βεβαίως πάντα γινόταν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας ε, και το αποτέλεσμα είναι ακόμη περισσότερος κατακαιρματισμός. Αν ε, δημιουργούμε μια πιο φτηνή και ευέλικτη αγορά εργασίας, ε, προσελκύει νέες θέσει εργασία και δημιουργείται νέος κατακαιρματισμός. Επίσης, κοιτάμε την οργάνωση αγορά εργασίας από τη Σκοπιά της σταδιοδρομίας. Ε, υπήρχε αυτό το θέμα εδώ και καιρό, αλλά τώρα το αγκαλιάζουμε και ακριβώς ε, περνάμε σε μια αρχή ευελιξία τη προσλήψη, αλλά βεβαίω αυτά τα οποία ακολουθούν, επενδύσει κτλ., αλλαγή σταδιοδρομία και το να πηγαίνουμε από τι πιο ευέλικτε στι πιο τακτικέ τα δουλειέ είναι αυτό το οποίο λείπει. Αλλά αυτό, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο πλαίσιο μια κρίση. Η τελευταία δεκαετία ήταν πολύ δύσκολη Οπότε αν ψάχνετε θαύματα στην αγορά εργασίας είναι δύσκολο αν δεν υπάρχουν νέες θέσει εργασίας, αλλά φαίνεται ότι σε πολλές χώρες αφήνω τις πιο προβληματικές. Φαίνεται ότι η οικονομία έχει περάσει τον κάβο και δημιουργούνται νέες θέσει εργασίας ε, στον ιδιωτικό τομέα. Thank you. Σας ευχαριστώ όλους, όλες και όλους για τις ε, παρεμβάσεις Έχουμε που και που κοινέ συνεδριάσει με άλλες επιτροπές, εμείς από την Επιτροπή Απασχόλησης, όπως τώρα με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Βλέπουμε λοιπόν τα θέματα συζήτησης, τα θέματα που απασχολούν. Έχουμε την κατάσταση της απασχόλησης, την κοινωνική κατάσταση, που είναι σημαντικά προβλήματα. Βλέπουμε τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για μια ακόμη φορά για τις παρεμβάσεις σας και νομίζω ότι μπορούμε εδώ να ολοκληρώσουμε αυτήν την συνεδρίαση λέγοντας ότι μπορεί να βρούμε τώρα μια πρόχειρη λύση, αλλά υπάρχει μέλλον.